Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας καλωσορίζω όλους στην Επιτροπή, αλλά και που μπορώ να καλωσορίζω τον Επιτροπό Αλμούνια για μια ανταλλαγή απόψεων. Έχω έναν ε, κατάλογο εδώ ε, των ε, επιτρόπων ε, που είχαμε υποδεχθεί, την Έλλη Κρούς το Σεπτέμβριο, τον Αλμούνια ε, με τους συντονιστές στις 4 Μαρτίου και η επόμενη συνάντηση μαζί σας θα είναι τον Οκτώβριο. Επομένως, ε, ήδη σας έχουμε δει αρκετά, θα σας ξαναδούμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα και θα σας δώσω το λόγο για 15 λεπτά περίπου και μετά θα, ακολουθήσουν, θα ακολουθήσει μια σειρά ερωταπαντήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα σε 15 λεπτά να σας ε, μιλήσω για κάποια στοιχεία τα οποία συνδέονται με την ε, ετήσια έκθεση ανταγωνισμού για το 2009 και να, σας, ε, και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου και κάποια σχόλια που αφορούν τον βασικό, τους βασικούς στόχους και τις δράσεις που αναλάβαμε τους τελευταίους μήνες. Από την τελευταία φορά που ήρθα εδώ, που ήταν η ακρόασή μου πριν ξεκινήσει η θητεία της νέας επιτροπής, έχουν συμβεί κάποια πράγματα. Από την ακρόαση επομένως, ε, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή οικονομικών θεμάτων. Είχαμε όμως ε, και κάποιες συναντήσεις ε, και συμφωνίες σε επίπεδο συντονιστών. Συνάντησα κάποιους από εσά ε, και αυτά τα οποία είχα πει και στην ακρόαση ότι θα είμαι πάντα ανοιχτό, έτσι ώστε να υπάρχει ένας ανοιχτό διάλογος μαζί σας και σαν Επιτροπή και μεμονωμένα δεν ήταν απλώς ένας ευσεβής πόθος. Είμαι πάντα στην διάθεσή σας για κάθε είδους διάλογο και ανταλλαγή απόψεων και είμαι έτοιμος να έρθω σε οποιαδήποτε κρεώση θεωρείται σκόπιμη. Καταρχάς, σας ασχοληθούμε λίγο με την ε, ετήσια έκθεση ανταγωνισμού για το 2009. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι λογικό η ουσία αυτής της έκθεσης να αφορά την οικονομική και την δημοσιονομική κρίση. Περιγράφει την ταχύτατη δράση που ανελήφθη από την Κομισιόν σύμφωνα με τους κανόνες για την κρατική ενίσχυση έτσι ώστε να προσφέρουμε έναν μηχανισμό για το συντονισμό των απαντήσεων των κρατών μελών στην κρίση και για να διευκολύνουμε ε, τα διάφορα μέτρα διάσωσης, να βοηθήσουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία χρειαζόντουσαν βοήθεια και αυτή η προσέγγιση πιστεύω ότι λειτουργήσε και λειτουργήσε αρκετά καλά θα έλεγα. Μας βοήθησε να αποφύγουμε την κατάρρευση του δημοσιονομικού μας συστήματος. Επίσης μας βοήθησε να αποφύγουμε αυτές τις κούρσες επιδοτήσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη, περιόρισε τις τρευλώσεις του ανταγωνισμού και περιόρισε και τα κίνητρα για την υπερβολική ανάλυψη κινδύνων. Επίσης ε, η δράση μας συνεισφέρει ε, οι τράπεζες ε, να αποκτήσουν μια πιο υγιή βάση εφόσον οι επιδοτήσεις οι οποίες δεν, δεν επιστρέφονται πρέπει να ενταχθούν σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης. Επίσης ε, εξασφαλίζουμε οι τράπεζες να πληρώσουν για τα λάθη του παρελθόντος και με τον τρόπο αυτό η Κομισιό λαμβάνει υπόψη και τον ηθικό κίνδυνο και ειλικρινά πιστεύω ότι είμαστε το μόνο δικαιοδοτικό όργανο το οποίο ρητά ασχολείται με τα θέματα ηθικού κινδύνου όταν ε, θέλουμε να υποστηρίξουμε το χρηματοοικονομικό σύστημα κατά διάρκεια της κρίσης. Από την, από την στιγμή που εγκρίναμε τα μέτρα διάσωσης ε, έχουμε σαν στόχο την μεσοπρόθεσμη, ε, μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και θέλουμε βέβαια, κοιτώντας μπροστά, να προχωρήσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και πώς θα γίνει η έξοδος από αυτή την κρίση. Όπως σας είπα και στην ακρόασή μου πριν από μερικούς μήνες, αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα, η έξοδος. Και η έξοδος τι σημαίνει. Σημαίνει δύο πράγματα. Καταρχάς σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε μέτρα του ανταγωνισμού έτσι ώστε να αποκτήσει ξανά η οικονομία, η μας μια δυναμική, να βοηθήσουμε τις οικονομίες μας να βγουν από την κρίση πιο ισχυρές και καλύτερα εξοπλισμένες για να αποκτήσουν μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα ότι οι τράπεζές μας ε, θα ε, προχωρήσουν σε μία αναδιάθρωση εφόσον είναι απαραίτητα απαραίτητο έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Τώρα, στον δημοσιονομικό και στο μη δημοσιονομικό τομέα της ε, οικονομίας μας θα πρέπει να ε, μην εξαρτώμεθα μόνο από την κρατική, να μην εξαρτώνται μόνο από την κρατική ενίσχυση οι τράπεζές μας. Δηλαδή, οι τράπεζες δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την κρατική υποστήριξη για περισσότερο χρόνο από ό,τι είναι απαραίτητο και θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από την αγορά. Η... Στο τελευταίο μας, στην τελευταία μας ανακοίνωση για την ε, εαρινή, αν θέλετε, ε, για τις το ενδεαρινό δελτίο για τις κρατικές ε, ενισχύσεις ε, έδειξε ότι μέχρι το τέλος του 2009 η χρήση των ε, κυβερνητικών εγγυήσεων περιορίστηκαν. Δηλαδή, στο πρώτο τρίμηνο του 2009 οι κυβερνητικέ ενισχύσεις αφορούσαν το 30% κατά μέσον όρων της συνολικής χρηματοδότησης των τραπεζών. Μέχρι το τέλο του έτου, το ποσοστό αυτό έχει πέσει στο 4%. Για να ενισχύσουμε αυτή την τάση, προσαρμόσαμε τους κανόνες όσον αφορά τις κρατικές εγγύησεις στον τραπεζικό τομέα. Από τον επόμενο μήνα, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2010, οι τράπεζες αυτές ε, που θα συνεχίσουν να ε, χρησιμοποιούν την ε, χρηματοδότηση θα αντιμετωπίσουν μια αύξηση όσον αφορά τα τέλη που θα στηρίζεται στην αξιοπιστία τους και στην φερεγγιότητά τους και οι τράπεζες που θα συνεχίσουν να εξαρτώνται στις ε, κρατικές ε, ε, ενισχύσεις επίσης θα πρέπει να υποβάλλονται σε μια αναθεώρηση βιωσιμότητας. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά την αγορά των κρατικών ομολόγων. Συνεργάζομαι πάρα πολύ στενά με τους συναδέλφους, τον κύριο Όλι Ρεν και τον Μισελ Μπαγνιέ, έτσι ώστε να διαχειριστούμε την έξοδο και την Τη στιγμή που θα γίνει αυτή η έξοδος χρειάζεται όμως ε, περισσότερο συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, μια κανονιστική μεταρρύθμιση έτσι ώστε να ε, γίνει η έξοδος αυτή με επιτυχία η πολιτική ανταγωνισμού έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτή τη κρίση. Όμω, η πολιτική ανταγωνισμού δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Και δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ο σωστό κανονισμό, η σωστή νομοθεσία και η πολιτική ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να χειραγωγηθεί έτσι ώστε να αντισταθμίσει την έλλειψη μια αποτελεσματική νομοθεσία. Τώρα, όσον αφορά την υποστήριξη που δίνουμε στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στο μη δημοσιονομικό σκέλο ε, τη ε, οικονομία, ε, τα μέτρα θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας αυτή την ύπαρξη του προσωρινού πλαισίου που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να, να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στην επίστοση και αυτό το προσωρινό πλαίσιο ε, πρόκειται να λήξει στο τέλος του 2010. Είναι πάρα πολύ νωρί ακόμα να ξέρουμε κατά πόσον χρειάζεται να παρατείνουμε την ισχύ αυτού του πλαισίου πέραν του 2010 και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε την αξιολόγηση αυτή το φθινόπωρο για να πάρουμε τι αποφάσει μα. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε ξεκινήσει μια διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και του ε, ενδιαφερομένου για την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου. Αυτή τη στιγμή ε, αξιολογούμε τι απαντήσει των κρατών μελών και των υπευθύνων, αλλά βέβαια δεν πρόκειται να σα ε, αποκαλύψω ένα μεγάλο μυστικό λέγοντα ότι οι απαντήσει είναι τελείω διαφορετικέ και αντιφατικές. Για μένα όμω είναι σαφή δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την ε, ε, φθήνουσα πορεία του, καθεστώτος, του εξαιρετικού καθεστώτος κρίσης και στον ε, δημοσιονομικό τομέα και στην πραγματική οικονομία. Όμως είναι σαφές επίσης ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν θα ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την, ε, τον οικονομικό τους δυναμισμό εάν στηριχθούν ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κρατική υποστήριξη. Γι' αυτό επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μπορέσουμε να δράσουμε γρήγορα και άμεσα όταν δούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Αλλά ούτω ή άλλως θα πρέπει να βγούμε με κάποιο τρόπο από αυτή την κρίση. Κάποιοι λένε βέβαια ότι οι κρατικέ ενισχύσει και η πειθαρχία όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει που επιβάλλουμε στις, ε, στην Ευρώπη καθιστά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, ε τις, τις καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικές και τις βάζει σε πιο δυσμενή θέση. Εγώ διαφωνώ. Οι κανόνες ε, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ε, προλαμβάνουν αυτές τις κούρσες επιδότησης ανάμεσα στα κράτη-μέλη, δημιουργούν ένα πλαίσιο ισότητας ε, για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και ενθαρρύνουν τις εταιρείες να είναι καινοτόμες, να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και να είναι υγιείς. Οι κανόνες ε, για τις κρατικές ενισχύσεις ενισχύουν και ε, τα κράτη-μέλη να προσφέρουν καλή βοήθεια. Δηλαδή, συνεισφέρουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ε, συνοχή, όπως παραδείγματο χάρη οι ενισχύσεις για τα project επενδύσεων σε, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή βοήθεια για επιχειρήσεις που δρούν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή ε, υποστηρίζουν, ε, αν θέλετε, ε, δημόσιες, στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία, ή διορθώνουν προβλήματα της, της αγοράς. Πιστεύω ότι αυτό του είδους η ενίσχυση θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική και θα ενθαρρύνει την ανάκαμψη. Ταυτόχρονα οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων αποθαρρύνουν τα κράτη-μέλη από το να προσφέρουν κακή ε, βοήθεια για να υποστηρίξουν ε, μη αποδοτικέ και μη ανταγωνιστικέ εταιρείε που αποτελούν ένα άχθο, ένα βάρο για, για, για τα δημόσια οικονομικά. Αυτό είναι, αποκτά μεγαλύτερη σημασία εφόσον τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να βρουν δημόσιες οικονομίε, αν θέλετε, για να περιορίσουν το, τα δημόσια ελλείμματα και το χρέος. Τώρα, ας δούμε τι γίνεται με το αντιτράστα και τις, με τους κανόνες αντιτράστα και με τις συγχωνεύσει. Το 2009 αντιμετωπίσαμε ε, κάποιες, ε, κάποιους οι οποίοι μας ζητούσαν, αντιμετωπίσαμε φωνές που μας ζητούσαν να περιορίσουμε κάπως την πολιτική για το αντιτράστα, να χαλαρώσουμε την πολιτική για το, για το αντιτράστα και τις ε, συγχωνεύσεις διότι είπανε ότι σε, σε περίοδο κρίσης θα πρέπει αυτοί οι κανόνες να χαλαρώσουν. Εγώ διαφωνώ απόλυτα, διότι πιστεύω ότι η, η, η συμπεριφορά ε, που παρεκκλίνει από μια σωστή πολιτική ανταγωνισμού και δημιουργεί καρτέλ ή ομίλου ή ε, οδηγεί σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πρόβλημα ε, και να, βλάψει τους καταναλωτέ επιτρέποντα τι εταιρείε να αυξήσουν τις τιμές τους. Εμείς ε, παραμένουμε στου κανόνες όσον αφορά τον έλεγχο των συγχωνεύσεων και ο στόχο μα είναι να δημιουργήσουμε ε, κανόν, παράγοντες ε, σωστού υγιούς ανταγωνισμού στην, στην αγορά. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε κάποιες εταιρείες, να αυξήσουμε τις τιμές. Κάτι τέτοιο θα κάνει την Ευρώπη λιγότερο ανταγωνιστική και γιατί θα αυξήσει τις τιμές. Όταν όμως ε, μια συγχώνευση δημιουργεί προβλήματα, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθούν ε, βιώσιμες διαρθρωτικές ε, λύσεις, έτσι ώστε να προστατεύσουμε και τους Ευρωπαίους καταναλωτές, που είναι και οι καταναλωτές αλλά και οι βιομηχανικοί καταναλωτές, όπως παραδείγματος χάρη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα θα πρέπει να δούμε ποιοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το βάρος της κρίσης. Ε, δεν πρέπει οι καταναλωτές να είναι αυτοί που θα αντιμετωπίσουν το βάρος της κρίσης. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία δεσποζουσών θέσεων. Έχουμε υιοθετήσει ε, αποφάσεις που αφορούν την απαγόρευση σχετικά με την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας με την Intel, Microsoft και Rambus και στον ενεργειακό τομέα. Ε, επίσης ανοίξαμε, ξεκινήσαμε κάποιες έρευνες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ε, όσον αφορά τις, ε, τα καρτέλ, έχουμε υιοθετήσει έξι αποφάσεις και έχουμε επιβάλει ε, κυρώσεις που ανέρχονται στο 1,62 δισεκατομμύρια ευρώ σε 43 εταιρείες. Πολλά από αυτά τα καρτέλ έχουν διεθνείς διαστάσεις, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία με τις, με τις αρχές ανταγωνισμού χωρών όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Ελβετία, Επίσης, ε, η, η έχει ασχοληθεί με μεγάλα καρτέλ που αφορούν παραγωγή, παραγω, παραγωγούς ε, ε μνήμης ε, που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές και στους σέρβερς Οι εταιρείες αυτές ε, πλήρωσαν κυρώσεις ε, ε, που ανέρχονται στα 331 εκατομμύρια και επίσης άλλες ε, υποθέσεις ελέγχονται. Τώρα, σαν αποτέλεσμα της κρίσης επίσης έχουμε και μια σημαντική μείωση στις απαιτήσει των εταιριών γιατί πολλές από αυτές τις εταιρείες δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τις κυρώσεις. Βέβαια, οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να ε, λειτουργούν αποθαρρυντικά. Ταυτόχρονα όμως ξέρουμε ότι δεν είμαστε εδώ για να επιβάλλουμε τους κανόνες ανταγωνισμού ε, παράλογα και να βγάλουμε από την αγορά κάποιες εταιρείες. Επομένως, οι εταιρείε ε, που μας ζητάνε ότι δεν, που μας ζητάνε δεν μπορούν να πληρώσουν, εξετάζουμε τα αιτήματά τους πάρα πολύ σημαντικά, σοβαρά και στην, ε, με τους άλλους επιτρόπους ε, το έχουμε συζητήσει. Προσπαθούμε να δούμε ε, πώς θα, θα υιοθετήσουμε μια συνεκτική ε, αντιμετώπιση για όλες τις εταιρείες ε, που μας λένε ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τις ποινές που τους έχουν επιβληθεί και θα πρέπει να, η, η, Κομισιόν εξετάζει την ρευστότητα, τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν οι εταιρείε, οι εταιρείε που δεν μπορούν να πληρώσουν τελικά θα δούνε τις κυρώσεις τους να μειώνονται ε, και να φτάσουν σε ένα επίπεδο όπου να μπορούν να τις πληρώσουν, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι αυτή ένα, μια θετική απάντηση ε, σε μια εταιρεία που μας λέει ότι δεν μπορεί να πληρώσει θα είναι κάτι το εξαιρετικό. Τώρα, πέραν της ε, κρίσης, μετά από την κρίση. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι διαδικασίες μας ε, θα είναι όσο δυνατόν καλύτερες και αποτελεσματικότερες. Όπως ξέρετε έγιναν πολλές ε, συζητήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες μας. Σε αυτές τις διαδικασίες και σε αυτές τις συζητήσεις έστρεψα την προσοχή μου, τις μελέτησα και κάτι τέτοιο θα συνεχίσουμε, διότι πιστεύω ότι το διοικητικό μας σύστημα στο οποίο η Κομισιόν έχει την ευθύνη να δρά σαν ένας αμερόληπτος και αντικειμενικός παράγοντας, έχει πολλές αρετές. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης, όμως οι θεμελιώδεις αξίες του συστήματός μας δεν θα πρέπει να αμφισβητηθούν. Τώρα, όσον αφορά τι ε, πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, έχουμε δύο πρωτοβουλίες ε, για το 2010 και το 2011. Ε, αυτές οι πρωτοβουλίες είναι καταρχάς μια αναθεώρηση για το, το θα αξιολογήσουμε τις οριζόντιες συμφωνίες συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνιών για την έρευνα και την ανάπτυξη και θα έχουμε μια συνάντηση με τους συντονιστές επόμενε εβδομάδες. Και το δεύτερο σημείο είναι το, η, η, η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει για τις ε, δράσεις όσον αφορά τις ζημιές. Έχουμε ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση και θα προσέξουμε ιδιαίτερα τις συμφωνίες που αφορούν την βελτίωση της καινοτομίας ε, και της ανταγωνιστικότητας ε, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μας και των ε, συμφωνιών, στάνταρ συμφωνιών. Τώρα όσον αφορά τις ε, ζημιές, πιστεύω ότι πριν εισάγουμε ένα σύστημα συλλογικής ανόρθωσης στην Ευρώπη θα πρέπει να σκεφτούμε ιδιαίτερα προσεκτικά. Και εγώ αλλά και άλλοι δύο συνάδελφο, ο συνάδελφοι, ο Τζον Ντάλι και η Βιβιέν Ρέντινγκ, ε, τα είπαμε αυτά και στις ακροάσεις μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Όπως βλέπουμε και από το αμερικανικό σύστημα, αυτή η συλλογική ανόρθωση μπορεί να οδηγήσει σε ένα σύστημα διαφορών Επομένω, Επομένως, αυτή... Και αυτό ξεπερνάει τον στόχο δηλαδή της ε, αντιστάθμισης της ζημιάς που υπέστη αυτός ο οποίος έχει βλαφθεί. Και επομένως αυτό το θέμα δεν συνδέεται μόνο με τον ανταγωνισμό. Γι' αυτό ακριβώς η Κομισιόν θα εξετάσει ε, πώς θα εισάγει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την συλλογική ανόρθωση. Πριν όμως αναλάβουμε οποιοδήποτε δράση θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τις κοινέ αρχές που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε, στους ε, διάφορους τομείς ε, προγραμματίζουμε με την Κομισιόν και με αυτούς τους δύο συναδέλφους που ανέφερα και προηγουμένως, Βιβιάν Ρέντιν και Τζον Τάλι, τον, ε, το φθινόπωρο να οργανώσουμε μια δημόσια διαβούλευση και μετά η Κομισιόν θα υιοθετήσει μια στάση, δηλαδή θα διαμορφώσουμε μία βάση για ε, μεμονωμένες νομοθετικές προτάσεις, όπως παραδείγματος χάρη οι δράσεις για, τις, για το αντιτράστο. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, πιστεύω, ότι έχουμε αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κρίσης. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα από, το, από την ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισμό. Καταρχάς εφαρμόσαμε ένα εξαιρετικό σύστημα, ε, πλαίσιο συγγνώμη, κρατικών ενισχύσεων, το οποίο βοήθησε ε, τις κυβερνήσεις να βρουν μια απάντηση στην κρίση. Έχουμε διαχειριστεί τις συνέπειες ε, της κρίσης αυτής στην οικονομία μας και δεύτερον έχουμε διατηρήσει ε, μια μια ισχυρή πολιτική ανταγωνισμού κάτω από δύσκολες συνθήκες. Επομένως, πιστεύουμε ότι θα είναι προς όφελον όλων των καταναλωτών της Ευρώπης να έχουμε μια ισχυρή ανταγωνιστική οικονομία. Thank you, I know you your Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ξέρω ότι θέλετε να πιείτε το καφέ σας που μάλλον θα έχει κρυώσει μέχρι τώρα. Άμα κρυγόρησα λέει ο Επίτροπος, όχι καλέ, έτσι το λέω. Τώρα θέλουν όλοι να σας ρωτήσουν και έχω τους εξής συναδέλφους και θα προτείνω τα εξής. Ένα λεπτό για ερωτήσεις και ε, μέχρι τρία λεπτά για τις απαντήσεις. Και αν ε, δεν είστε καλά παιδιά θα αρχίσω να σας επιπλήττω. Λοιπόν, να σας διαβάσω το κατάλογο, ξέρετε πού είστε. Darlene McCarthy, Sanchez Sophie Andreas Schwab, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Liam Huangot, Annie Podimata, Vicky Ford, Thomas Mann, Jürgen Klute, Ramon Tremosa. Udo, you wanted to come in there possibly. Θέλετε ενδεχομένω να ζητήσετε το λόγο. Α, είπατε. Έχω 120 ερωτήσεις εγώ. Αλλά επειδή εκπροσωπείται η πολιτική μου ομάδα πολύ ωραία, ο συνάδελφος Πίτερ Σίμεν ίσως και δεν χρειάζεται να γραφτώ κι εγώ σήμερα. Ωραία. Ferreira, uh, Ωραία. Ο Ούντο είπε ότι δεν θέλει να πάρει το λόγο. Ζων Πολ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρα. Αγαπητέ Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την τόσο λεπτομερή παρουσίαση που έδειξε όλα τα βασικά προβλήματα που σας απασχόλησαν φέτος και θα συνεχίσουν να σας απασχολούν και ευχαριστώ που πήρατε υπόψη σας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες, οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις. Ένα θέμα είναι οι κυρώσεις μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών ανάμεσα στις εταιρείε. Ε, η θέση σας έχει εξελιχθεί ή πιστεύετε ότι η βάση για τον υπολογισμό της ε, ποινή ε, πρέπει να, να είναι η μητρική εταιρεία και όχι η εταιρεία που έκανε το σφάλμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ένα άλλο θέμα με το οποίο δεν, δεν ασχοληθήκατε, αλλά μπορεί να είναι καινούριο και δεν θέλω άμεση απάντηση, αλλά στην πολιτική ανταγωνισμού που αφορά τον γεωργικό τομέα. Ποια είναι η άποψή σας. Ξέρετε ότι η μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ ε, βρίσκεται εν εξελίξη, ακόμα το σκεφτόμαστε το θέμα και τίθενται κάποια συγκεκριμένα θέματα ε, και κάποια ερωτήματα στον γεωργικό κόσμο όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Η μεταφορά των κανόνων ανταγωνισμού για τις κλασικές επιχειρήσεις στον γεωργικό τομέα μπορεί να είναι δύσκολη. Επομένως, ε, ε, ήθελα να ξέρω αν έχετε ξεκινήσει την σκέψη για αυτό τον τομέα. Δεν χρειάζεται να μου δώσετε μια απάντηση τώρα, διότι πιστεύω ότι μάλλον σε εμβριακή φάση βρίσκεται η σκέψη σας. Προτιμώ να απαντήσω άμεσα μετά από κάθε ερώτηση, δηλαδή να δίνω και την απάντηση. Με βάση τον, η βάση, σαν βάση υπολογισμού των κυρώσεων ε, εφαρμόζουμε τα ίδια κριτήρια τα οποία βρίσκονται και στους προσανατολισμούς του 2006. Δηλαδή έχουμε τα ίδια κριτήρια, το μόνο το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι με την κρίση έχουμε περισσότερες αιτήσει ε, για inability to pay, δηλαδή αδυναμία πληρωμής ε, και είμαστε υποχρεωμένοι να ε, προχωρήσουμε με την ανάλυση που, έκανα και στην, που έδωσε και στην παρουσία μου, παρουσίασή μου. Τώρα, για το δεύτερο θέμα που θίξατε, συζητάμε την πολιτική ανταγωνισμού και τη γεωργική πολιτική. Το συζητάμε και γενικά και πιο συγκεκριμένα όταν η ομάδα υψηλού ε, επίπεδου για το γάλα ε, ε, υπέβαλε τα απορίσματά της την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, έχει σαν στόχο να, να συγκλίνει την λειτουργία των γεωργικών αγορών με τις κανονικές αγορές. Επομένως δεν θα πρέπει να αποσύρουμε την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού Πιστεύω ότι αυτό που είναι απαραίτητο είναι να προσαρμόσουμε τους κανόνες ανταγωνισμού στις ιδιαιτερότητες των γεωργικών προϊόντων. Παραδείγματος χάρη ε, για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Συζήτησα και με τον Γάλλο Υπουργό Γεωργίας και του είπε ότι θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες πολιτικής ανταγωνισμού αλλά υπάρχουν κάποια παραδείγματα. <coughs> Π.χ. ας πούμε εμείς έχουμε, θέλουμε να ενημερώσουμε τον τομέα για τα παραδείγματα προβλήματα που υπάρχουν σε πολλές χώρες όπου παραδείγματο χάρη έχει οργανωθεί η συζήτηση για τις τιμές των γεωργικών προϊόντων με έναν πολύ πιο λογικό και αποτελεσματικό για τα συμφέροντα των παραγωγών τρόπο. Ε, και αυτό σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα σε κάποιο τομέα. Υπάρχουν ε, υφιστάμενα προβλήματα του τομέα για τα οποία χρειάζεται μια πολιτική απάντηση, δηλαδή την εφαρμογή μια κατάλληλη πολιτικής, αλλά δεν είναι θέμα πολιτικής ανταγωνισμού. Παραδείγματο χάρη σε ορισμένου γεωργικού τομεί, αυτό που χρειάζεται είναι μια καλύτερη οργάνωση, μια καλύτερη ένταξη των διαφόρων ε, σταδίων παραγωγής ε, έτσι, ώστε, να μπορούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν διαπραγματεύσεις να έχουν την ε, κατάλληλη ικανότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ιδέα της αναδιάρθρωσης, ε, αλλά είπατε για να μην υπάρχουν επικίνδυνες συμπεριφορέ, είπατε να υπάρχουν πληρωμές στα μερίσματα, για να υπάρχουν ε, κρατικές ε, ενισχύσεις. Οι περισσότεροι κατανοούν γιατί συνέβη ό,τι συνέβη, όμως μήπως είναι κατά του, αντι, του ανταγωνισμού αυτά τα μέτρα, το ότι θα πρέπει οι εταιρείε να εξακολουθούν να πληρώνουν τεράστια τεράστιους μισθούς και τεράστια μπόνους. Θα θέλα να με ενημερώσετε για, την διεύρυνση, για τη διερεύνηση της κατάχρησης θέσεως στα ασφάλιστρα ε, τα CDS ε, και επειδή μας είχατε πει ότι θα ληφθούν κάποια μέτρα το 2010, ε, θα συνεχιστούν τα μέτρα αυτά το 2011, το 2012 ή θα είναι SAE. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί ούτω ή άλλω να αντιμετωπιστεί ε, μέσω ε, των μέτρων και το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στην ανάλυση της κατάστασης των τραπεζών αλλά ως ε, τμήμα που ε, ε, ως τμήμα ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να δούμε την κατάσταση στον τραπεζικό τομέα όχι μόνο βάσει των συνεπειών στο ευρύτερο σύστημα που το γνωρίζουμε τους τελευταίους μήνες αλλά υπάρχουν και κάποια ζητήματα διοντολογίας και υπάρχουν και κάποια πολιτικά προβλήματα που υπησέρχονται σε αυτήν ε, την, σε τους υπερβολικούς ε, μισθούς και που δεν έχουν καμία σχέση με τα αποτελέσματα ε, της εταιρεία. Εξακολουθούμε βέβαια να προσέχουμε πολύ, να δίνουμε προσοχή στα ζητήματα αυτά. Και όσον αφορά τις δεσμεύσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα βλέπουμε ε, κατά πόσο οι ε, υποχρεώσεις τους και ε, η πληρωμή των υπερβολικών αυτών μισθών αντίκειται στο, στη, στην, στην ευρύτερη κατάσταση του ανταγωνισμού. Προσέχουμε λοιπόν με πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα τι συμβαίνει στον τομέα αυτό ε, όχι μόνο ε, ως ε, αρμόδια για τον ανταγωνισμό αλλά και ο Μισελ Μπαρνιέου, είναι μου, ασχολείται με το ζήτημα αυτό και επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το τι συμβαίνει. Όσον αφορά την Ιρλανδία, όπως και σε άλλα κράτη-μέλη, Λαμβάνουμε αιτήματα για την παράταση των σχεδίων εγγυήσεων που εγκρίθηκαν στην αρχή της κρίσης και όπως είπα και στην παρουσίασή μου, Έχουμε κάποιους ε, όρους ε, εγγύηση των τιμών σε περίπτωση που τα χαμηλότερα επιτόκια είχαν ε, ως αποτέλεσμα καλύτερες συνθήκες ε, ε, σε σχέση με χρηματοπιστωτικά συστήματα που μπορεί να επιβίωναν καλύτερα λόγω της θέσης τους στην αγορά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, τα προβλήματα, ότι οι προβληματικές τράπεζες θα λάβουν μεγαλύτερη ενίσχυση από τις ε, τράπεζες ε, που δεν ε, αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα. Εμείς αναλύουμε τις συνθήκες και αναλόγως αποφασίζουμε κατά πόσο μπορούμε να παρατείνουμε τα μέτρα που εγκρίναμε στην αρχή. Αν τα κράτη-μέλη μας ζητήσουν περαιτέρω παράταση, εμείς μπορεί να δώσουμε μία παράταση για έξι μήνες, αυτή, αυτός είναι ο γενικός κανόνας, αλλά για την περίπτωση της Ιρλανδίας το Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους, συγγνώμη, του προηγούμενου έτους, όταν στην αρχή της κρίσης αποφασίστηκαν κάποια μέτρα, θα ε, αναθεωρηθεί τώρα κατά πόσο αυτή η απεριόριστη εγγύηση, αυτές οι απεριόριστες εγγύησεις ε, θα διακοπούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, για την οικονομική κατάσταση Μιλήσατε για τη σταδιακή έξοδο από την κρίση, το phasing out, ε, όσο εξομαλύνεται η κατάσταση αυτό να εκπνέει. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αρκετή διαφάνεια αυτή τη στιγμή, γιατί και οι ενισχύσει χρειάζονται διαφάνεια πάντα. Στη συνέχεια, για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η η πολιτική ανταγωνισμού έχει εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται και σε σύγκριση και σε σχέση με τη στρατηγική 2020, με την οικονομική πολιτική μπορεί να αποδώσει και τέλος το θέμα των καταναλωτών. Μιλήσατε για οριζόντια εξέταση, για να έχετε μια συνολική εικόνα και μετά με μονομενα μέτρα. Έχετε χρονοδιάγραμμα. και για κάποια νομοθετική πρωτοβουλία για το φθινόπωρο. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση στα ισπανικά. Διαφάνεια στις ενισχύσει. Μα καταρχήν ε, με διαφανή τρόπο χορηγούνται. Τουλάχιστον κάθε φορά που μεμονωμένα ε, έχουμε απέναντί μας ε, μια χρηματοπιστωτική οντότητα. Το σχέδιο διάσωσης, αναδιάρθρωσης, βιωσιμότητας, κάθε φορά ζητούμε τις προφορίες. Οι τράπεζες, ας πούμε, με τις οποίες συναλλασσόμαστε κάθε φορά, μας στέλνουν ε, όλες τις προφορίες, ορισμένες αντιστέκονται, αλλά εμείς επιμένουμε και τελικά είναι υποχρεωμένες. Αλλιώς δεν είναι θετική η απόφαση στο σχέδιο επιβίωσής τους και διάσωσης. Ε, λοιπόν, μιλάμε για μεμονωμένη αντιμετώπιση και εκεί υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Και είναι πολύ θετικό αυτό που υποστήριξε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόσφατα. Δηλαδή, πριν να αρχίσουμε να μιλάμε για αναδιάρθρωση μεμονωμένων τραπεζών ή κρίση, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια απέναντι στην αγορά. Και έχουμε αυτά τα τεστ αντοχής, stress test, που θα ε, δημοσιευθούν τις επόμενες ε, εβδομάδες. Είναι μια άριστη πρακτική. Στη συνέχεια, πολιτική ανταγωνισμού ανάκαμψης οικονομίας. Αναφέρθηκα στις κρατικές ενισχύσεις, τις καλές και τις κακές, εντός αγωγικών πάντα, στο κείμενο. Όταν κάποιος διαβάζει ένα κείμενο, καμιά φορά υπάρχουν εισαγωγικά που δεν φαίνονται. Ε, καλές και κακές εντός εισαγωγικών. Ποιες είναι οι καλές ενισχύσεις. Θα πρέπει ε, όσο γίνεται περισσότερο να τις διακρίνουμε ε, και να είμαστε λεπτοί στην προσέγγιση μας, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο στον προϋπολογισμό του κάθε κράτους να επιλέγουμε προτεραιότητες και εργαλεία για να χρησιμοποιούνται τα δημόσια κονδύλια στην υπηρεσία της στήριξης περιφερειών πιο απομακρυσμένων, στην απασχόληση, στις ε, επενδύσεις για καινοτομία, κεφάλαιο κινδύνου, εκπαίδευση, παιδεία, ε, με μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι στο παρελθόν. Και δική μας πλέον ευθύνη που ε, πρέπει να ελέγχουμε τις δημόσιες ενισχύσεις είναι να είμαστε πιο αυστηροί στις αρνητικές μας αποφάσεις και να ε, δηλώνουμε, ε, να κηρύσουμε μάλλον μη συμβατές με τη συνθήκη ε, εκείνες τις προτεραιότητες που δεν εγγράφονται στη στρατηγική 2020 και τις αντίστοιχες ενισχύσεις. Και δική μας ευθύνη λοιπόν δεν είναι μόνο να λαμβάνουμε συγκεκριμένες αποφάσεις αλλά και να ενημερώνουμε όλους τους φορείς, ιδιώτες και δημόσιο, ποιο είναι το πλαίσιο των αποφασιών μας και όσο χρειάζεται να ενημερώνονται, να βελτιώνονται οι προσανατολισμοί όπου βασίζουμε τις αποφάσεις μας και θα το πράξουμε αυτό στο μέλλον. Και τρίτη ερώτηση ε, για την οριζόντια δημόσια διαβούλευση για όλες τις συλλογικέ δράσεις θα γίνει όντως το φθινόπωρο. Υπολογίζω, χωρίς να δεσμεύομαι τώρα για συγκεκριμένη ημερομηνία, ότι αρχές του 2011 ε, βάσει αυτής της διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταλήξει σε συμπεράσματα και τη στιγμή που θα βγάλει αυτά τα οριζόντια συμπεράσματα για συλλογικέ δράσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεμαι να υποβάλω ε, στο Σώμα των Επιτρόπων και ε, στη συνέχεια στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την προετοιμασία ε, της αποζημίωσης από βλάβες που προκύπτουν από στρεβλώσεις ανταγωνισμού. Η Σοφή Νετφελτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε στην πρώτη σας ε, συνάντηση με την Επιτροπή μας. Ω εισηγήτρια για την ε, περσινή έκθεση έχω πολλά ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα Κυρίως μεθοδολογικής φύσεως είπατε κατά την ακρόαση σας και το επιβεβαιώσατε και στην ομιλία σας ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς εγκρίναμε το Μάρτιο με τεράστια πλειοψηφία ε, ένα ψήφισμα για την προηγούμενη έκθεση με πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και συγκεκριμένα αιτήματα και θα ήμασταν πολύ ευγνώμονες αν μπορούσατε να μας απαντήσετε ειδικότερα κατά προτίμηση εγγράφος για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα αιτήματά μας και τα ερωτήματά μας. Δεύτερον, αν δω την ε, φετινή έκθεση, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι μία σύνοψη δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της, της ασματικότητας, που είναι ένα ερώτημα που θέσαμε στην περσινή έκθεση. Θέλουμε να ξέρουμε τα αποτελέσματα όλων των μέτρων, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε αν είναι αποτελεσματικέ οι πολιτικέ μα. Ξέρουμε ότι αυτό είναι αποκλειστικό, είναι τομέα αρμοδιότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ξέρω ότι έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, αλλά εγώ σε συγκέντρια, θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα παραπάνω, αλλιώ δεν έχει νόημα να συζητούμε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Κυρία Πρόεδρε, αυτό νομίζω που θέλουμε να ξέρουμε είναι την αποτελεσματικότητα και τα ενδεχόμενα στρεβλωτικά, ε, τις στρεβλωτικές συνέπειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως επίσης και το προσωρινό, ε, τα αποτελέσματα του προσωρινού πλαισίου ε, ενίσχυσης. Όπως είπαμε και στο ψήφισμα μας, ε, τα στοιχεία που έχουν ε, διαθέσει τα κράτη-μέλη θα τα χρησιμοποιήσετε ως βάση για την απόφαση του ναι ή όχι, θα του, του αν θα αποφασίσετε την παράταση ή όχι των μέτρων. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται και μία ανεξάρτητη ανάλυση όλων αυτών. Τελευταίο ερώτημα. Ζητήσαμε κάναμε και κάποια ερωτήματα ανατομέα και θα ήθελα να ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα λάβει υπόψη τη και αν ε, όχι, για ποιο λόγο. Απάντηση. Για το πρώτο ερώτημά σας, ναι, θα αποστείλω απάντηση γραπτός ε, σε κάθε ένα από τα ερωτήματα που θέσατε για το 2008. Ε, έχω ένα πολύ καλό έγγραφο ε, στα, στο φάκελό μου και θα ήταν πολύ εύκολο να το μετατρέψω σε επιστολή προς την Επιτροπή σας. Όσον αφορά τώρα την έκθεση του 2009, μα, με ρωτήσατε για ποιο λόγο δεν, ε, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Γιατί, κοιτάξτε, δεν έχουμε ε, ολοκληρώσει τη χρήση όλων αυτών των μέσων. Είμαστε στη μέση ε, των ε, μέσων αυτών που αποφασίσαμε στην αρχή της κρίσης. Ενδεχομένως να είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δυστυχώς είναι πολύ νωρίς να προβούμε σε αξιολόγηση του πώς έχουμε χρησιμοποιήσει τα επιπλέον αυτά μέτρα. Όσον αφορά τώρα τις τρευλωτικές συνέπειες της κρατικής ενίσχυσης. Κοιτάξτε, δεν θα βασίσω, ούτε θα προτείνω στους συναδέλφους να βασίσουν την απόφασή τους ε, για τη σταδιακή έξοδο από αυτό το καθεστώς και στο, χρηματοπιστωτικό, και στο μη χρηματοπιστωτικό τομέα, μόνο βάσει των απαντήσεων που λαμβάνουμε. Για τους λόγους που είμαι σίγουρος ότι θα κατανοήσετε, αν ρωτήσω, όταν ρωτάω τα κράτη-μέλη, πιστεύετε ότι αυτό το εξαιρετικό καθεστώς πρέπει να συνεχίσει τα μισά λένε ναι και τα άλλα μισά κράτη-μέλη λένε όχι. Όταν εγώ συναντώ, όπως σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, με ε, οργανισμούς εργοδοτών από κράτη-μέλη που λένε παρακαλούμε διατηρήστε 100% το προσωρινό αυτό καθεστώς ε, ενώ άλλοι λένε ότι ε, δεν επιθυμούν αυτό το καθεστώς. Τι να σας πω, στερεοφωνικά δηλαδή ακούω διαφορετικές ε, ε απόψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει το, ο τίτλος της ε, απάντησής μας δεν θα βασιστεί σε ερωτήσεις που θέτουμε προς τα κράτη-μέλη. Και στο τρίτο ερώτημά σας θα ήθελα να απαντήσω ότι υπάρχουν χρήσιμα μέτρα που δεν μπορούν εκ των προτέρων να ανακοινωθούν, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των φαρμακευτικών, γιατί χρειαζόταν μια διερεύνηση επιτόπου και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση των αρμοδιοτήτων μας για διερεύνηση τριών-τεσσάρων τομέων, να χρησιμοποιούμε δηλαδή ανθρώπινους σπόρους σε τομείς χωρί να είμαστε βέβαιοι για την προστιθέμενη αξία. Πρέπει να επικεντρώνουμε τι προσπάθειέ μα σε τομεί προστιθέμενη αξία ε, και για του καταναλωτέ. Αν εκ των προτέρων εμείς ανακοινώνουμε ότι θα αρχίσουμε συγκεκριμένες τομεακές έρευνες, ενδεχομένω, να μην έχουμε τελικά ε, πάρα, πολλά, πάρα, πολύ, πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά ε, στην διερεύνησή μας, στην έρευνά μας. Ähm, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να πω καταρχάς ότι ως αρμόδιος για τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς κύριε Επίτροπε, είστε σε πολύ καλύτερη θέση να εξηγείτε τα μέτρα από ότι στο παρελθόν. Γι' αυτό θεωρώ τόσο σημαντικό όταν είμαστε σε χαλεπούς καιρούς οικονομικά να τηρούμε το δίκαιο του ανταγωνισμού και την πολιτική των ενισχύσεων. Για να το καταφέρουμε όμως θα πρέπει να εξηγούμε σωστά την πολιτική μας και θέλω αυτό να το τονίσω πραγματικά. Την περασμένη εβδομάδα δηλώσατε ότι δεν απαιτούνται ε, τραπεζικές εγγυήσεις ε, σε περίπτωση καταβολής προστήμων και κυρώσεων, επιβολής κυρώσεων και από το 2008 στην έκθεση του ανταγωνισμού λέγεται ότι για ε, επιχειρήσεις ενός ε, προϊόντος μόνο product ε, businesses θα έχετε ειδικά μέτρα. Το ρώτησε προηγουμένως και ο κύριος Κοζές. Εμείς πάντα μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς θα λέτε τώρα αυτά μόνο product businesses. θα υπάρχει έκτακτη ρύθμιση εκεί. Στη συνέχεια, ε, της δαπάνης προσωπικού, εγώ ήμουν εισηγητής για τον προϋπολογισμό και θέλουμε να υποστηρίξουμε τη δική σας γενική διεύθυνση για να γίνεται μια καθαρή ανάλυση της αγοράς και μας είπαν όμως ότι υπάρχει αρκετό προσωπικό εκεί. Οπότε νομίζω ότι μπορείτε να αποκριθείτε και στα όσα ζήτησε η κυρία Ινετφέλτ. Και ένα τελευταίο προσπαθεί η Πρόεδρος να με ανακαλέσει την τάξη, να μου θυμίσει τον χρόνο. Υπάρχει ένα απομεινάρι από την έκθεση του 2008 η χάρτα του θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να μπει στη, Λισαβόνα, στη νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Από το 2003 το συζητάμε αυτό. Γιατί υπάρχουν ζητήματα ιδιοκτησίας, κυριότητας ε, των ε, ε, επιχειρήσεων που δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμα. Εκκρεμεί αυτή η ιστορία. Τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή, η Πρόεδρος. Συγγνώμη, που σας ε, λέω να βιαστείτε, αλλά και όσοι θα πάρουν το λόγο πιο μετά πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα να εκφραστούν όσο με όσου πήραν ε, το λόγο στην αρχή. Να απαντήσω στα ισπανικά. Καταρχάς συμφωνώ μαζί σα. Ακριβώ σε τέτοιου χαλεπούς καιρού από πλευρά οικονομική, κοινωνική, μέχρι και πολιτική. είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε, να εξηγούμε και να εξηγούμε κάθε φορά τι κάνουμε, για ποιο λόγο το κάνουμε και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουμε. Αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω μεταξύ άλλων. Αν μετρούσα τις διασκέψεις ή τις δημόσιες εμφανίσεις μου από τότε που ανέλαβα αυτό το χαρτοφυλάκιο το Φεβρουάριο, θα έβγαιναν πάνω από μία την εβδομάδα. Δημόσιες εμφανίσεις ομιλώ, πέρα από ε, τέτοιου είδους συνεδριάσεις και είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Για ε, τις επιχειρήσεις ενός προϊόντος, που συνήθως είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πράγματι, δίνω προσοχή και μελετώ πώς ε, λειτουργεί η εφαρμογή των σημερινών προσανατολισμών ως προς τα πρόστιμα, ε, πώς αυτό επιδρά στις εταιρείες και στο ισολογισμό τους. Έχω την υπόθεση τύραμς υπόψη μου που λύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μετά από συμφωνία. Πώς το λένε αυτό, settlement. Στα ισπανικά δεν ξέρω, διακανονισμός πάντως είναι τις επόμενες εβδομάδες θα ε, λάβουμε και άλλες τέτοιες αποφάσεις και θα διδαχθούμε από την εμπειρία και κάποια στιγμή θα κάνουμε το ίδιο που κάνουμε σήμερα για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν αδυναμία πληρωμών. Δηλαδή, ακόμα περισσότερο θα ε, έχουμε τελειοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε τα πρόστιμα. Τώρα όταν ε, δηλώνω αδυναμία πληρωμών ε, δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ καλά στον υπολογισμό, αλλά δεν το ξεχνάω. Για την προσωπική ερώτηση και το θέμα του προσωπικού για τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμό, όταν έρθει στο Κοινοβούλιο ο κύριος Σεύκοβιτς, συνάδελφός μου αρμόδιος για ε, το ε, ανθρώπινο δυναμικό, του ανθρώπινου πόρου να του το πείτε. Δημόσια δεν θέλω να ζητήσω περισσότερου πόρου για τη γενική διεύθυνσή μου, διότι αν δημόσια βγαίνει ο κάθε επίτροπο, θα είναι παραφωνία. Ε, αν το πείτε εσεί καλύτερα. Ξέρετε έχετε καλύτερα επιχειρήματα από μένα για να τα εξηγείτε αυτά τα θέματα, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερου ανθρώπινου πόρου. Και για την τελευταία ερώτηση, αν κατάλαβα καλά αυτό που με ρωτάτε, είναι τι γίνεται με την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού μετά από την κύρωση της Ιθήκης Λισαβόνας και, την, και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ενσωματώνεται στο βασικό πρωτογενές δίκαιο. Και είναι η νομολογία του Δικαστήριου του Στρασβούργου. Εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά εκ πρώτης όψης δεν φαντάζομαι να έχει αυτό μεγάλη εμβέλεια επιπτώσεις. Ειλικρινά σας το λέω. Αλλά θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε γιατί έχει τη σημασία του.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 Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Πίτροπε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπουμε. Νομίζω ότι αυτός ο διάλογος είναι πολύ χρήσιμος. Μία παρατήρηση σχετικά με αυτά που ο Ζων Πολ Γκοζές. Όταν λέτε ότι στον γεωργικό τομέα δεν τίθεται υπαμφισβήτηση ο ανταγωνισμός. Ο, συμφωνώ. Όμως ο ανταγωνισμός θα πρέπει να μας βοηθήσει έτσι ώστε οι αγοραστές να είναι περισσότεροι. Και εδώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Όταν υπάρχει μια τέτοια συγκέντρωση σε επίπεδο αγοραστών δεν είμαι σίγουρη ότι έχουμε, μια ελεύθερη, έχουμε έναν ελεύθερο ανταγωνισμό. Επί της ουσίας, μια και θέλετε γραπτά να βλέπετε τα πράγματα. Θα σας υποβάλουμε και γραπτά την ερώτησή μας με την Σοφή. Βέβαια, υπάρχει ένα μια φήμη και δεν, ξέρω, δεν νομίζω ότι είσαστε εδώ για να σχολιάσετε τις φήμες, αλλά τέλος πάντων, όταν μιλάμε για κάποιες συμφωνίες, ε, τότε θα πρέπει να ξεκινάμε και κάποιες έρευνες. Υπάρχουν, ε, ακούγεται ότι υπάρχει μια συνάντηση στη Νέα Υόρκη κάποιων που θέλουν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των νομισμα, του νομίσματός μας. Ε, μήπως θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει κάτι το παράνομο Επομένως η Κομισιόν θα έπρεπε να κάνει μια μικρή έρευνα διότι αυτέ είναι, αυτές είναι συμπεριφορέ ε, τις οποίες δεν εκτιμάμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Γκουλάρ, όταν απάντησαν ε, στον συνάδελφό σας, τον κύριο Γκοσές, είπα ε, αναφέρθηκαν μάλλον στα αιτήματα τα οποία πήραμε από το γεωργικό τομέα. ξέρω ότι έχετε δίκιο ότι Προφανώς θα πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά του κατά πόσον υπάρχουν προβλήματα από πλευρά των αγοραστών, δηλαδή από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Εγώ όμως αναφερόμουν στα αιτήματα τα οποία έχουμε πάρει από τους παραγωγούς και υπάρχουν και κάποιες δημοσιεύσεις επίσημες της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που δείχνουν ακριβώς ποια είναι τα περιθώρια τα οποία ε, έχουν ε, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις διαπραγματεύσεις από πλευράς των παραγωγών. Δεν είναι κείμενα βέβαια νομοθετικού περιεχομένου, δεν έχουν νομική ισχύ, είναι ενημερωτικά έγγραφα που δίνουν τα περιθώρια τα διαπραγματευτικά που έχουν παραγωγή. Και βέβαια από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να αγνοούμε τι συμβαίνει και από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Βέβαια, με κάποιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού είδαμε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις τις οποίες παρακολουθούν. Ακόμα όμως, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, δεν, ούτε στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ούτε τώρα, δεν υπάρχουν ε, αποδείξεις που να μας αναγκάζουν να ξεκινήσουμε μια έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε όμως σε εβδομαδιαία επαφή με τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού που ασχολούνται με το θέμα. Τώρα, για το δεύτερο θέμα. Α, ποιο ήταν αυτό. Ναι, όντως, έχετε... αλήθεια είναι. Το συζήτησα το θέμα με τις Αμερικανικές Αρχές. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε αυτού του είδους τις συναντήσεις να τις ε, συγκρίνουμε ε, με τις ε, οδηγίες που δίνουμε για τα δημοσιονομικά εμείς. Αυτό όμως δεν είναι η άποψη του ενός εμπειρογνώμονα. Παίρνοντας το καπέλο τώρα του τι τις θέσεις που είχα πριν ως προηγούμενος επίτροπος, το να σας πω ότι, να, ότι πιστεύω ότι ένα δείπνο μπορεί να θίξει το, το ευρώ, δεν το πιστεύω αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες σύντομες ερωτήσεις για τις κρατικές εγγύησεις. Ε, αναγνωρίζετε προφανώς ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δεν ε, είσαστε όμως πολύ συγκεκριμένος ε, για το πώς θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε τις κάποιες στρεβλώσεις αγοράς που δημιουργούν αυτές οι ενισχύσεις προς την τράπεζα. Δεύτερο αυτό. Και τι γίνεται με τις στρεβλωτικές συνέπειες που θα είχε αυτή η ενίσχυση που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις Εθνικές Τράπεζες. Επίσης για τα ανθρακοριχεία ε, θα συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έρευνα και αν ναι Επίσης δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει μια έρευνα αγοράς για την, ε, για την διανομή, για τα σούπερ μάρκετ κλπ. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει και κάποια... Ε, κάποια συμφωνία ανάμεσα στους, στο λιανεμπόριο Επίσης, τι γίνεται με τη στρέβλωση ανταγωνισμού που μπορεί να δημιουργήσουν κάποιες φορολογικέ διατάξεις που υιοθετούν τα κράτη-μέλη. Τώρα, για τις κρατικές εγγύσει, απαντάει ο κ. Σαλμούνια και για τις ε, στρεβλωτικές συνέπειες που μπορεί να έχουν. Όπως ξέρετε, υιοθετήσαμε τέλος του 2008, αρχέ του 2009, κάποιους προσανατολισμούς για τις τιμές και για τις συνθήκες των ε, ε, χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σαν, σαν έκτακτη εγγύηση για την κρίση. Αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται για, την, για κάθε μεμονωμένη ανάλυση των εθνικών προβλημάτων και αν υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο δεν συνάδει με τις γενικούς προσανατολισμούς που συζητήσαμε και υιοθετήσαμε, τους το λέμε ότι για να εγκριθεί το εθνικό πρόγραμμα θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις και να προσαρμοστεί το πρόγραμμα στις, στους γενικούς προσανατολισμούς και το ίδιο γίνεται και για κάθε μεμονωμένη περίπτωση την οποία να αναλύουμε. Ήδη έχουμε υιοθετήσει μεμονωμένες αποφάσεις για πολλές περιπτώσεις. Έχουμε όμως ακόμα 40 περιπτώσεις ατομικών ε, μεμονωμένων υποθέσεων όπου θα πρέπει να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις από μόνους μήνες. Για τον άνθρακα. Δεν γίνεται μια έρευνα. Αυτό το οποίο προετοιμάζουμε είναι ένας κανονισμός για τις ε, κρατικές ενισχύσεις που δίδονται στον άνθρακα. Θα υποβάλουμε αυτό το σχέδιο κανονισμού, πρόκειται για ένα ε, κανονισμό του Συμβουλίου. Θα το, θα υποβάλουμε σε δύο εβδομάδες και προβλέπεται νομίζω για την ε, συνάντηση των Επιτρόπων της 6ης Ιουλίου και μετά αφού υιοθετηθεί το σχέδιο κανονισμού και θα ακολουθηθεί όλη η διαδικασία των συζητήσεων ο κανονισμός αυτός απαιτεί την ομοφωνία του Συμβουλίου και το Κοινοβούλιο έχει, έχει κάποια θέση εδώ. Δεν ξέρω ποια ακριβώ θέση έχει. Νομίζω ότι θα πρέπει να γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο πριν ε, υιοθετήσει οριστική άποψη το Συμβούλιο. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσω για το τι θα γίνει. Τώρα για τη μεγάλη διανομή, για τους μεγάλους για τους διανομής. Δεν είπα ότι δεν θέλω να γίνει μια έρευνα. Είπα ότι απλώς δεν θέλω να, να εξαγγείλω εξάντε κάποιες έρευνες που ε, απαιτούν και ε, φυσική παρουσία στους χώρους των επιχειρήσεων που θα αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας. Διότι δεν θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η έρευνα, για να το πω με κομψό τρόπο. Δηλαδή να εξαγγείλουμε εξάντε ότι θα κάνουμε μια έρευνα σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Όχι βέβαια ακόμα κατά τη διάρκεια της θητείας μου δεν έχουμε ξεκινήσει τομεακές έρευνες. Θα τις κάνουμε όμως γιατί στο παρελθόν είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα αυτών των ε, ερευνών. Τώρα για τα θέματα τα φορολογικά, για τους φόρους, ε, το συζητήσαμε διμερώς ε, πλιστάκης. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις. Υπάρχει μία νομολογία, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την οποία να μπορούμε να συζητήσουμε με όλο το συμβασμό με τα δικαστήρια, που λέει ότι εφόσον ο φόρος είναι ο ίδιος σε κάθε ένα από τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να δεχτούμε ότι το επίπεδο φορολόγησης μπορεί να είναι διαφορετικό εκτός ε, για τους ε, φόρους που είναι εναρμονισμένοι στα διάφορα κράτη-μέλη. Τώρα είναι λογικό αυτό ή δεν είναι, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι όταν εφόσον έχουμε μια εσωτερική αγορά δεν είναι απόλυτα λογική η ρίση αυτή. Αλλά αυτά λέει η νομολογία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στη διένεξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και Γαλλίας σε ό,τι αφορά τους γαλλικούς σιδηροδρόμους ζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει το καθεστώς της SNCF με την πρόφαση ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της ε, ήταν στρέβλωση του ανταγωνισμού όταν ζητούσε δάνεια από τις τράπεζες. Εκεί βρήκα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβολικά μαξιμαλιστική στην ερμηνεία της, υπερβολική ως προς τα κείμενα ε, όταν ε, γίνεται λόγος για τη διάνοιξη του ανταγωνισμού. Δεν επιβάλλει αλλαγή του καθεστώτος ή του κανονισμού της εταιρεία. Και δεν σημαίνει ότι ε, το να ανοίξει στον ανταγωνισμό μια εταιρεία ίσον ιδιωτικοποιείται, έτσι δεν είναι. Θα ήθελα να σας πω επίσης και να θυμίσω ότι κρατικές εγγύησεις για τις δημόσιες επιχειρήσει. Ε, δικαιολογούνται γιατί δεν είναι επιχειρήσεις που έχουν ίδια κεφάλαια όπως οι ιδιωτικέ εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Άρα για να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας που έχουν ο κοινοφελή, θα πρέπει να έχουν και κρατικές ενισχύσεις. Για να είναι λοιπόν αποτελεσματική και να βαθμολογεί, θα πρέπει να βαθμολογείται ε, μια εταιρεία. Αυτό δεν με σοκάρει ο σοσιαλιστή, ούτε τον Κοζέ, το φίλο μου που είναι εγκολικό. Μάλλον σοκάρει μόνο του φιλελεύθερου. Μπορείτε να μα διαβεβαιώσετε ότι δεν θα ξανάρθει ε, στην αντεπίθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πού ε, είναι η σκέψη και ο προβληματισμό σα για την οδηγία των κοινοφιλών υπηρεσιών που μα είχε τάξει ο κύριος Μπαρός Μίλησα ε, μια μισή-δύο ώρες ε, στο κοινοβούλιο, ε, σε μια διπλανή αίθουσα για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Σιμών ήταν εκεί και μπορεί να σας περιγράψει τι είπα. Και νομίζω ότι ήμουν σαφής όσον αφορά τις δηλώσεις στα θέματα αρχής και για το πώς θα εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές. Τώρα βέβαια είναι και αυτή είναι μια συζήτηση που μπορούμε να επαναλάβουμε εδώ, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερο από πέντε λεπτά. Τώρα για το θέμα της SNCF. Η Κομισιόν δεν, άλλαξε, δεν ζήτησε αλλαγή του καταστατικού, κύριε Βουλευτά. Δεν το ζητήσαμε. Και είναι ένα δημόσιο έγγραφο, διότι δημοσιο... δημοσιεύθηκε στον τύπο. Ε, διέρευσε στον τύπο. Το έμαθα εγώ από τον τύπο και το διάβασα και είδα ε, την επιστολή. Δεν ζητήσαμε αλλαγή του καταστατικού δεν πήραμε καμία θέση επί του καταστατικού, επί της θέσης. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι είναι ή τι θα πρέπει να είναι μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση. Είμαστε ουδέτεροι σε αυτό το θέμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η στρέβλωση του ανταγωνισμού. Για να φέρει ο κύριος Λαμπέρ, εάν υπάρχουν ε, επιχειρήσεις ε, για τις οποίες εγγυάται ένα κράτος και κάποιες άλλες επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει κρατική εγγύηση, εκεί όντως υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Και η Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Γαλλίας ε, ε, ε, πήρε, λήφθη μια απόφαση στο Γαλλικό Κοινοβούλιο να αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και Θέλω να ξέρω με τους υποστηρικτές αυτής της φιλελευθεροποίησης, έτσι όπως ζητάτε τώρα, απαιτείτε τώρα, τι θα γίνει. Ζητάτε μια θέση όσον αφορά τις κρατικές εγγύσεις. Αυτό γίνεται. Εφόσον πρόκειται για μια ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού τομέα ή του δημόσιου τομέα, μπορεί οποιοδήποτε στην Ισπανία, στη χώρα μου, έχουμε ιδιωτικές, ε, ιδιωτικές τράπεζες, τα ταμιευτήρια, τα οποία δεν, είναι, ε, δεν έχουν το καθεστώς δημόσιας εταιρείας, αλλά βέβαια ο καθένας μπορεί να τις χαρακτηρίσει όπως θέλει, αλλά πάνω μέσα στην αγορά χρειάζεται μια ισότητα. γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με τις δημόσιες υπηρεσίες που θέλουμε να προσφέρουμε και στους καταναλωτές μέσω αυτών των επιχειρήσεων. Ιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. I think that you will need your translation Δύο σύντομε ερωτήσει θέλω να κάνω. Η πρώτη αφορά στη λειτουργία των οίκων αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα σημεία στα οποία έχει εστιαστεί η κριτική ε, αφορά στο γεγονός ότι οι υπηρεσία αξιολόγηση υπάρχει υπερσυγκέντρωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περιορισμένο δηλαδή αριθμό εταιριών, με έδρα μάλιστα εκτός τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κύριο λόγο, γεγονός που εγείρει σημαντικά προβλήματα ανταγωνισμού. Ήθελα να σα ρωτήσω κατά πόσο έχετε πραγματοποιήσει έρευνα ε, για να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις της ε, υπερσυγκέντρωσης των υπηρεσιών αξιολόγησης στην ευρωπαϊκή ένωση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις αυτό είναι το ένα και το δεύτερο αφορά σε αυτά που μας είπατε για τους κανόνες αντιτράστ και τις συγχωνεύσεις τα προβλήματα ρευστότητας που παρουσιάζονται στο τραπεζικό τομέα σε ορισμένες χώρες είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε εξαγορές και σε συγχωνεύσεις τραπεζών αυξάνοντας τα προβλήματα ε, μονοπωλιακής πρακτικής σε αυτές τις περιπτώσεις και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή είναι μια εξέλιξη που σας ανησυχεί και αν μπορούν να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για τους οίκους αξιολόγησης rating πιστοληπτικής ικανότητας, αυτό που κάνουμε εμείς είναι βάζουμε μια τάξη, ρυθμίζουμε. Έχω την αίσθηση ότι κυριαρχεί η γενική ρύθμιση παρά η αναπερίπτωση ρύθμιση ε, που ήταν ε, στην προηγούμενη θητεία και της Κομισιόν και του Κοινοβούλιου. Υπήρξε ένας πρώτος κανονισμός που έβαζε όρους για μητρώα, για διαφάνεια, για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κτλ. Και πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ε, υποβάλει εν ευθέτω χρόνο μετά την ε, συζήτηση που θα πρέπει να γίνει ένα ευρωπαϊκό οργανισμό ή μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση αυτών των οίκων αξιολόγησης αυτό είναι ο σωστός δρόμος. Και δεν νομίζω ότι είναι αμυγός πρόβλημα ανταγωνισμού αυτού. Έχουν μακρά ιστορία σφαλμάτων, κακών πρακτικών, στρεβλών καταστάσεων αυτές οι ε, εταιρείε και οι οίκοι. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, είναι θέμα ανικανότητας βασικά και ε, για ε, τις τραπεζικές ε, καμιά φορά χρειάζονται. Η ε, συγχώνευση βοηθάει για να βελτιωθεί στην ανασυγκρότηση ένα τραπεζικό ίδρυμα. Εδώ, σε αυτή τη χώρα, είναι γνωστή μια περίπτωση συγχώνευσης τράπεζας που χρειάστηκε. Αλλά, ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών θα πρέπει να ανησυχούμε από μονοπωλιακές πρακτικές. Έχουμε άλλα στοιχεία για να ανησυχούμε για το πώς λειτουργούν οι χρηματαγορές, το σύστημα ολόκληρο, αλλά τα μονοπόλια όχι, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτός ο κίνδυνος είναι στη συγκέντρωση μεγάλων τραπεζών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εκεί μπορούμε να το δούμε. Λίγες τράπεζες που πολύ γρήγορα έγιναν ακόμα λιγότερες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στην Ευρώπη αυτό το stress test που μόλις έχει ε, ανακοινωθεί είναι 25 τράπεζες. Δεν είναι μόνο 25 οι τράπεζες, εκατοντάδες είναι στην Ευρώπη, 25 είναι οι μεγαλύτερες. Και σε πολλα κρατημέλη κράτη-μέλη μας τα επόμενα χρόνια ε, ακριβώς για καλύτερες υπηρεσίες και πιο αποτελεσματικές μπορούμε να δούμε συγχωνεύσεις τραπεζών χωρίς να θεωρώ ότι υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι στιγμής κίνδυνοι εκεί κατάχρηση δεσπόσα θέση ή μονοπωλιακές πρακτικές. Άλλα προβλήματα υπάρχουν πολύ σοβαρά που θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε, αλλά αυτό το μονοπώλιο δεν νομίζω. Βίκη. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε, πάρα πολύ ωραίο είναι που συνδέσατε την ανάπτυξη με τον ε, ανταγωνισμό με την πολιτική ανταγωνισμό, όπως επίσης ε, και η κατανόηση και η ευαισθησία σας ε, ως προς το ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις για την ανάπτυξη και ότι τα εμπόδια προς την επένδυση είναι κάτι το οποίο σε όλες τις πολιτικές ομάδες συμφωνούμε. Ε, αφορά πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα, ε, τα ε, equities ε, και τα, τη δυνατότητα εγγραφής των τραπεζών σε αυτές, στα equities. Ήθελα να σας ρωτήσω αν δεν υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός σε αυτήν την αγορά. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι παίκτες στην αγορά αυτή. Και ένα ακόμη ερώτημα και το έθεσα ως ε, νέο ε, μέλος ε, την, το περασμένο φθινόπωρο. Τι γίνεται με τα πρόστιμα Φαντάζομαι ότι μένουν σε λογαριασμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που τα λαμβάνετε ε, και κάποια στιγμή μετά τα επιστρέφετε στα κράτη-μέλη. Μέχρι, στιγμής, μέχρι τη στιγμή που θα τα λάβουν όμω πίσω έχουν ξεχάσει για ποιο ακριβώ σκοπό είχαν επιβληθεί τα πρόστιμα αυτά. Μήπω θα μπορούσατε λοιπόν να, ε, να βρεθεί ένα τρόπο ε, τα χρήματα αυτά να επιστρέφονται νωρίτερα ναι, θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να ε, υπάρχουν καταρχάς. Θα αρχίσω από τη δεύτερη ερώτηση. Όταν ε, είναι υπό έφεση το πρόστιμο που έχει επιβληθεί, πρέπει να περιμένουμε μην τυχόν μειώσει το πρόστιμο ή λάβει μια διαφορετική απόφαση το δικαστήριο και μήπω τυχόν επιστραφεί ένα τμήμα του ποσού ή όλο το ποσό στην εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι αν συμφωνήσει το δικαστήριο με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν υπάρχει έφεση, ε, τότε ε, πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα. Βέβαια θα ήθελα να παραμείνουν και κάποια χρήματα εδώ γιατί η περισσότερη δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται αλλά οι κανόνες είναι κανόνες. Όσον αφορά το ερώτημα το άλλο που μου θέσατε θα προσπαθήσω να το διερευνήσω να διερευνήσω τι ακριβώς κάνουν ε, οι Βρετανικές αρχές Έχουμε κρεμίσει υποθέσεις, ε, γνωρίζετε ότι υπήρχαν κάποιες υποθέσεις και εξακολουθούν να υπάρχουν εκρεμείς υποθέσεις για τα MIF, τα multilateral, ε, Intervention Fees σε συνεργασία με τη Mastercard και τη Visa. Συμφωνήσαμε για τις πιστοτικές κάρτες. Ε, ε, έχουμε ήδη κάποιες συζητήσεις και με τη Visa αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε έτσι όλα τα προβλήματα ε, που έχουμε ε, με κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή η μεταφορά χρημάτων. Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο από άποψη ανταγωνισμού αλλά από κοινού με τον Μισελ Μπαρνιέ κατά τα ερχόμενα έτη είναι τα ΣΕΠΑ. Το, είναι το ΣΕΠΑ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών. Αυτό πρέπει να το επιτύχουμε. Και έχω αποστείλει επιστολή στον Μισελ Μπαρνιέ και απάντησε αμέσως θετικά συνεργαζόμαστε για το θέμα αυτό για να προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο αυτό το σύστημα ευρωπαϊκών πληρωμών ε, δεν έχει ακόμη ε, λειτουργήσει, πώς μπορούμε να υπερβούμε τα εμπόδια. Είναι ένα ζήτημα ανταγωνισμού, είναι ένα ζήτημα ε, ρύθμιση. Σε μερικές περιπτώσεις η αυτορύθμιση είναι λίγο προχωρημένη και δεν είναι ο συντομότερος δρόμος για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε συνεπώς το επεξεργαζόμαστε. Ε, το ζήτημα το οποίο αναφέρατε δεν αφορά καταρχάς ε, αποκλειστικά το σύστημα πληρωμών. Είναι γεγονό όμω ότι στο πλαίσιο του τραπεζικού τομέα είναι πολύ ενδιαφέρον. Σε μερικέ περιπτώσει ε, επαφίεται ε, στου φορεί ανταγωνισμού, σε άλλε περιπτώσει είναι ένα ζήτημα προστασία των καταναλωτών ε, και πολλέ αρχέ αρμόδιε για τον ανταγωνισμό ε, σε κρατικό επίπεδο ασχολούνται με το ζήτημα αυτό σε εθνικό επίπεδο γιατί ακριβώ δεν είναι διασυνοριακό το σύστημα. Αν όμω προχωρήσουμε προ ένα πραγματικό ε, σύστημα πληρωμών θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπίζονται πολλά από αυτά τα ζητήματα. Έχω και εγώ μια σύντομη ερώτηση. Επτά ακόμη συνάδελφοι θέλουν να σας θέσουν ερωτήσεις και έχουμε ακόμη δέκα λεπτά. Πιστεύετε ότι μπορούμε να τους ακούσουμε. Σε ομάδες θα τους ε, ακούσουμε. Τόμας Μαν. Ε, κύριε Πίτροπε, Ευχαριστώ πολύ. Σε πολλούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ζήσαμε το γεγονό ότι δεν μα ακολούθησαν οι πολίτε. Ανοίξαμε μια ομπρέλα για προστασία και μα προσάπτουν ότι είναι για τι μεγάλε εταιρείε, για τι τράπεζε και οι μικρομεσαίε είναι εκτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η συγχωνεύση των τραπεζών δεν είναι ζήτημα. Αλλά επειδή υπάρχει αδιαφάνεια εκεί και δεν μπορεί κανεί να διακρίνει ποια είναι τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που κυκλοφορούν και υπάρχουν, ερωτώ, τι ε, μέτρα έχετε για την ανθιάθρωση των τραπεζών οι ε, τράπεζες ε, που διαθέτουν όλα τα προϊόντα επιτρέπεται ακόμα να λειτουργούν έτσι μια τράπεζα να διαθέτει τα πάντα ή θα το περιορίσετε αυτό και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι υπουργοί οικονομικών συνεδριάζουν ε, Σαββατοκυριακό άρον άρον βιάζονται προσπαθούν να βρουν αποτελέσματα αυτό δεν είναι σαφής εικόνα δεν θα μπορούσε να βγει μια τριανδρία και να πει εγώ είμαι αρμόδιος για τον ανταγωνισμό και ο Ρεν που τον ξέρω πολύ καλά και έχει ένα χαρτοφυλάκιο που το ξέρω κι εγώ και ο Μισελ Μπαρνιέ που μόλις ε, το χαρακτηρίσατε ΣΕΡΠΑ να προετοιμάσετε λοιπόν την οικονομική διακυβέρνηση και να ε, σας ελέγχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι άρον άρον. Ε, ευχαριστώ. κύριε Αλμούνια, θέλω να επανέλθω στην πρώτη ερώτηση της κυρίας Ποδηματά για τους οίκους αξιολόγησης, της πιστοληπτικής ε, ικανότητα. Είπατε ότι δεν είναι πρόβλημα ανταγωνισμού, αλλά πρόβλημα ανικανότητα. Δεν μου φτάνει αυτή η απάντηση, δεν μου αρκεί ακριβώ. Τρει ουσιαστικά είναι οι οίκοι αυτοί που κυριαρχούν στην αγορά. Ο λιγοπόλιο είναι καμία σχέση με ανταγωνισμό, η μικρή μόνο και η μεθοδολογία τους είναι γνωστή στον τύπο ότι είναι όλα πάρα πολύ θολά, συγκεχημένα, σκοτεινά, προβληματικά. Έχουν όμως πολύ μεγάλη ε, δύναμη και επηρεάζουν ε, και τη θέση ολοκλήρων εταιριών ή και οργανισμών. Και όντω είναι πρόβλημα ανταγωνισμού για μένα και θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό. Και σε σχέση και με την αξιολόγηση κρατών ή κρατικών δανείων. Και επειδή είναι έτσι όπως είναι η ε, αγορά, δεν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να το καταργήσει τελείως αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα με ενδιαφέρει πολύ η θέση σας. Καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Η οικονομική ιστορία μας διδάσκει ότι για να βγούμε από χρηματοοικονομική κρίση ε, η πρώτη προτεραιότητα και προϋπόθεση είναι να εξηγιαθεί το χρηματοοικονομικό σύστημα ε, ξανάρχεται ρευστό και κεφάλαιο στην τράπεζα και ανακάμπτει η οικονομία στην Ευρώπη, δυστυχώ στην Ισπανία όχι. Για το 2010 η Κεντρική Τράπεζα της χώρας σημειώνει μείωση της διοδότησης και των οικογενειών και των επιχειρήσεων. Γιατί λοιπόν η Ισπανία δεν επέλεξε ένα σύστημα που έχουν ακολουθήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες για να εξηγιάνουν τις τράπεζες. Το σύστημα της Bad Bank, μια κακή τράπεζα που καθαρίζει από τα τοξικά ε, στοιχεία ενεργητικού της τράπεζε και απορροφά ε, τις απώλειες. Στην Ισπανία το ΦΡΟΠ που είναι το Ταμείο Αναδιάρθρωσης έχει ε, μεγάλο επιτόκιο ε, σε χαμηλό διάστημα και δεν απορροφά τις απώλειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έπρεπε να είχε πέμβει εκεί πιο ενεργά και δραστήρια για να φτιάξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα εξηγήσεις των τραπεζών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να απαντήσω στον κύριο Μαν. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει ένα δόγμα για το τι τράπεζες θα πρέπει να υπάρχουν, καθολικών υπηρεσιών, λιανικής, επενδυτικές, χωριστές τράπεζες. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό οικονομικό πολιτισμό, κουλτούρα, δομή, διάρθρωση, απαιτήσει, ανάγκες διαφορετικές. Προηγούμενα, εγώ δεν τολμώ να μπω σε αυτά τα χωράφια. Αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι όλοι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και τα ιδρύματα θα πρέπει ε, να τη πολύ καλή ρύθμιση και πάρα πολύ καλή εποπτεία. και οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να τη χάνουν τις ιδιαίτερες προσοχές όχι μόνο του εποπτικού συστήματος αλλά να υπάρχουν και εκείνοι οι κανόνες συνετού διαχείριση για να μην αναλαμβάνουν κίνδυνο περισσότερο από εκείνο που μπορούν να καλύψουν και να χρηματοδοτήσουν. Αυτές είναι βασικές αρχές. Από εκεί και πέρα ε, εφαρμόζονται διαφορετικά στις τράπεζες που έχουν καθολικές υπηρεσίες, που είναι επενδυτικέ, που ε, ε, είναι τράπεζες που ε, χρηματοδοτούν επιχειρήσεις κτλ. Για την Τριανδρία τώρα και στην προηγούμενη θητεία και σε τούτη εδώ, οι τρεις αρμόδιοι επίτροποι για οικονομικά και νομισματικά, για εσωτερική αγορά και ανταγωνισμό και ε, ο πρόεδρος μαζί και το ιδιαίτερο γραφείο του, έχουμε ουσιαστικά καθημερινό συντονισμό καμιά φορά σε επίπεδο επιτρόπων, καμιά φορά σε επίπεδο διευθυντών ε, των γραφείων μας ή μεταξύ των υπηρεσιών. Πάντως συντονισμός υπάρχει και είναι απαραίτητο και σχεδόν καθημερινός. Το να το ονομάσουμε τώρα οικονομική κυβέρνηση, αυτό θα γεννήσει μεγάλους φθόνους ε, και ζήλιες σε άλλα θεσμικά όργανα, όχι σε τούτο. Ε, για το rating ε, έκανα ένα λογοπαίγνιο γιατί στα ισπανικά ο ανταγωνισμός είναι κομπετένσια και η ανικανότητα είναι incompetencia. Ε, ε, το θέμα λοιπόν είναι ότι χρειάζεται περισσότερη ρύθμιση. Αυτή είναι η ουσία. Και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ρυθμίσει στοιχεία των εικοναξιολόγησης ορισμένα και με πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα θητεία θα έχετε και άλλα στοιχεία να ρυθμίσετε. Και είναι ανάγκη αυτό όντω. Το rating τώρα η αξιολόγηση των δημοσίων χρεών ή κρατών. Εγώ έχω την άποψή μου γι' αυτό. Αν είναι σκόπιμο ή όχι να χαρακτηρίζουν ε, κρατικά ομόλογα. Έχω άποψη, δεν θα την πω δημόσια, αλλά την έχω. Ε, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος αν μπορούμε να αποφύγουμε ακριβώς οι αγορές που αγοράζουν το χρέος και διαπραγματεύονται για το χρέος και στο πρωτογενή και στο δευτερογενή κλάδο της αγοράς. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο εμπιστεύονται αυτούς που αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα, τη φερεγγιότητα κτλ. των κρατικών ε, χρεογράφων κάθε κράτους. Υπάρχουν πρωτοβουλίες, υπάρχουν ιδέες που ακούγονται πάρα πολύ καλές και πρόσφορες για το πόσο ε, θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ε, υπολογισμού του κινδύνου για τα κρατικά χρέη. Αλλά ας μην γελιόμαστε οι αγορέ θα εμπιστεύονται εκείνου που εκείνου θεωρούν αξιόπιστο. Και υπάρχουν ε, τελικά πραγματικότητες που δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Και ο κύριος Τρεμόσα, πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μα είπε, αλλά θα πρέπει να συζητηθούν στην Ισπανική Βουλή, όχι εδώ. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ τι να σα πω, ε, αναλύουμε το κάσο τη Ισπανία, Φιλανδία, Ιρλανδίας, τη Λετωνία, κάθε κράτο ξεχωριστά. Για το πώς ε, σώζει κάθε χώρα τις τράπεζες, πώς τις ε, ενισχύει, αν αυτό συνάδει με τις κρατικές ενισχύσεις και όπως αυτές έχουν οριστεί ε, για την εφαρμογή του σε περίοδο κρίσης, όπως τις περιγράψαμε και τις εγκρίναμε στις τέσσερις σχετικές ανακοινώσεις από το φθινόπωρο του 2008 μέχρι τα μέσα του 2009. Αυτό αφορά και την Ισπανία και οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τελευταίοι τέσσερις ομιλητές, όλοι μαζί. Η κυρία Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίσαμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα clearing system ε, των ε, τραπεζών που χρεοκοπούν. Ε, Το πρόβλημα είναι ότι η κρίση άφησε τις τράπεζες, τα κράτη και τους πολίτες πολύ πιο αβέβαιους και ανήσυχους για τον κίνδυνο ευρωπαϊκών φορέων που ξεφεύγουν κάπως από τον ελεγχό μας. Αυτό το πρόβλημα της έλλειψης εμπιστοσύνης νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μήπως μπορείτε να μας πείτε για αυτά τα μέτρα ανάπτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών οργάνων και πώς μπορούμε να διασκεδάσουμε αυτούς τους φόρους ότι τα πάντα θα είναι πλέον ε, υπό την αρμοδιότητα τεράστιων επιχειρήσεων. Το κόστος για τις τράπεζες μήπως τελικά θα μετακυλιστεί στην ε, πραγματική οικονομία. Και κάτι ακόμη. Η κρίση μας άφησε κάποιους πιο αδύναμους και κάποιους ισχυρότερους. Η πολιτική ανταγωνισμού θα προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όταν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι πλέον πολύ μεγάλες, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα ε, από τις δημοσιονομικές ε, χρηματοοικονομικές αγορές να περάσουμε στις ενεργειακές αγορές. Θέλετε, ε, θέλετε και το κάνετε εδώ και χρόνια να εφαρμόσετε κανόνες ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας. Υπάρχει μια νέα διαφορά που παρουσιάστηκε στους ε, συνεργάτες, στους συνεταίρους αν θέλει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, ε, ανάμεσα στην Ρωσία και στην Λευκορωσία, όχι ανάμεσα στην Ρωσία και στην Ουκρανία αυτή τη φορά. Μία χώρα όμως, η Λιθουανία, δεν παίρνει ε, πλέον φυσικό αέριο, διότι βασικός προμηθευτής της είναι από την Λευκορωσία. Εδώ υπάρχει, είναι μια απόδειξη έλλειψης παντελούς ανταγωνισμού στην, ε, στον ενεργειακό τομέα. Η Κομισιό τι θα πρέπει να κάνει ή εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται. Ο κύριος Σίμων. Χωρίς μικρόφωνο όμως δυστυχώς. Ευχαριστώ. Στο συγγνώμη. Ευχαριστώ που ήρθατε και χθε ε, στο Intergroup για τις δημόσιες υπηρεσίε και μιλήσατε πραγματικά για τις αντισταθμιστικές ε, πληρωμές σε τρίτους από τα κράτη για την ανάληψη υπηρεσιών κοινοφελειών. Σύντομα μόνο μιλήσατε για την έρθιμη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε την εξή αντίφαση, αντιπαλότητα. Από πλευράς τοπικών αρχών οτά δηλαδή των κρατών μελών ακούμε ότι με τα πρωτόκολλα που αφορούν τις ΔΕΚΟ ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε μια σχετικοποίηση του δικαίου ανταγωνισμού ότι, μπορούν, ότι έχουν το δικαίωμα οι δήμοι και οι κοινότητες ε, να διοργανώνουν και να επομίζονται αυτές τις υπηρεσίες και μάλιστα ενισχύεται αυτό το δικαίωμά τους. Στις δικές σας υπηρεσίες ε, ε, Όμω τονίζουν ότι το δίκαιο ανταγωνισμού είναι δίκαιο ανταγωνισμού, το τονίζουν τρει και τέσσερι φορέ και τελεία και δεν αλλάζει τίποτα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Εσεί αυτό πώ το ερμηνεύετε, αυτό το, την ένταση που δημιουργείται, γιατί είναι πεπισμένη τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση ότι έχει βγει ενισχυμένη. Και το άρθρο 14 τη Ειδίκης Λισαβόνα δίνει τη δυνατότητα σε νομοθεσία πλαίσιο, πάντα στι 10, ε, και ανοίγει το ενδεχόμενο πολλών ερμηνεών. Η δική μου ομάδα πάγια ε, έχει ένα αίτημα σχετικά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ρυθμιστεί ε, κλαδικά ή ορισμένοι δεν θέλουν καθόλου ρύθμιση. Και κάποια συνεργάτη σας είπε «Α, μα καλά, έτσι δίνανται λέει, μόνο σάλ γράφει, δεν σημαίνει ότι είναι και υποχρεωτικό». Αυτό το είπε δική σας συνεργάτη, η κυρία Κράτσα υποχρεωτικο αυτο το ειπε δικη σας συνεργατη κυρια κρατσα παρακαλω Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, σε πρόσφατη συνέντευξή σα, αναφερθήκατε στο ενδεχόμενο να υπάρχει ένα νέος κύκλος στήριξη τραπεζών. Ε, κυρίως νομίζω ότι αναφερθήκατε και σε δύο περιπτώσεις ε, των χωρών, την Ελλάδα και την Ισπανία ε, παράλληλα έχουμε και τη διαδικασία stress test η οποία φαίνεται ότι θα υιοθετηθεί. Ε, πώς θα συνδυαστούν αυτά τα δύο, θα περιμένετε το τεστ για να δείτε ε, ποιες, που υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι για να υπάρξει η διαδικασία διάσωσης. Και δεύτερον θα σας πω πώς αυτό συνδέεται με τον ανταγωνισμό. Μήπως υπάρξουν ε, αντιδράσεις από τις τράπεζες ή από χώρες που δεν θα είναι μέσα σε αυτό το νέο κύκλο στήριξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Φερέιρα πρώτα. Συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχει ανάγκη στην Ευρώπη να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο επίλυσης ε, ε, της κρίσης. Από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν το έχουμε. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν κάποιους μηχανισμούς αποτελεσματικούς επίλυσης κρίσεων για τους δικούς τους οργανισμούς κάθε φορά. Ε, διαφέρουν τα εργαλεία από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένα κράτη δεν υπάρχουν καν ε, αρκετά αποτελεσματικά τέτοια εργαλεία και στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις εμείς μέσα από τη χρήση των κρατικών ενισχύσεων και τον τρόπο με τον οποίο τις ρυθμίζουμε και με την ανάλυση των προγραμμάτων διάσωσης που κάνουμε και των σχεδίων αναδιάρθρωσης, εμείς λοιπόν δρούμε ως τέτοιο ε, ίδρυμα επίλυσης διαφορών. Ένα έγγραφο πρόσφατα δημοσίευσαν γνωστοί οικονομολόγοι που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ευρώπη και διερωτώνται μήπως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ανταγωνισμό θα έπρεπε να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός τέτοιος οργανισμός. Εγώ δεν θα φτάσω μέχρι εκεί, απλώς διαπιστώνω ότι ε, ε, έτσι έχει η κατάσταση, δεν είναι η καλύτερη δυνατή και θα πρέπει κάπως να σκεφτούμε τι να κάνουμε εκεί. Ένα δεύτερο στοιχείο με το οποίο συμφωνώ απολύτως, τα εξή δύο. Υπάρχει μια πρόκληση και όχι μόνο στην Ευρώπη πώς θα ρυθμίσουμε και θα παρακολουθούμε και θα υποπτεύουμε τις ε, ε, εταιρείε ή τους οργανισμούς που έχουν συστημικό κίνδυνο, too big to fail δηλαδή, με τρόπο που να μην είναι εκ του ασφαλούς ε, κάποιοι διευθυντές ή στελέχοι όταν έχουν πρόβλημα θα τους σώσει το κράτος εις βάρος της τσέπης του φορολογουμένου γιατί δεν μπορούν να τους αφήσει να αναβαγίσουν. Αυτό θα πρέπει να περιοριστεί όσο γίνεται. Και μετά συμφωνώ απολύτω με αυτό που λέτε ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, σωστή κατανομή του φόρτου, ένα burden sharing, δίκαιη. Ε, προσπαθούμε εμείς να ε, προωθήσουμε την δίκαιη κατανομή ε, των θυσιών και των βαρών που χρειάζονται για την αναθεάθρωση των τραπεζών και αυτές οι προσπάθειες δεν θα πρέπει να πέφτουν μόνο στους ώμους. Καμιά φορά δυστυχώς είναι ε, αναπόφευκτο αυτό εν μέρη να πέσουν στους ώμους των φορολογουμένων, αλλά γιατί όχι και εκείνοι που συνεισφέρουν στην κατάσταση αυτή, στους αρμόδιους διαχειριστές ε, των οργανισμών αυτών, στους ε, μετόχους, στο βαθμό του δυνατού και στους πιστωτές και αν μπορεί αυτό να το ζητήσει κάποιος. γιατί αυτό μπορεί να έχει ανεπιθύμητες ε, συνέπειες, ε, δηλαδή να, πρέπει οι πιστωτές να έρθουν να βοηθήσουν στη διάσωση μιας τράπεζας, γιατί μπορεί μετά να μην θέλουν να τους λεφτά. Και είναι άλλο πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει οπωσδήποτε όμως λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλιώς ε, το διστοτικό μας σύστημα δεν θα έχει τις απαραίτητες άμυνες, τα αντισώματα, για να μην πέσουμε στην ίδια κατάσταση που είδαμε από το 2007 και μετά. Τι γίνεται τώρα με το φυσικό αέριο που με ρωτήσατε. Σε ορισμένα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε φορά που η Ρωσία ή η Λευκορωσία έχουν προβλήματα και μεταξύ τους ή η Ουκρανία, αυτό δεν είναι θέμα ανταγωνισμού καταρχήν. Είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας. Στη συζήτηση που είχαμε αυτά τα χρόνια, κάπως προχωρήσαμε, αλλά όχι αρκετά. Πριν από λίγο καιρό είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια συζήτηση που έγινε στο Κοινοβούλιο για μια πρόταση που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με Εθνικά Κοινοβούλια για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Ενέργειας. Βέβαια αυτό χρειάζεται αλλαγές στη συνθήκη κτλ. Χωρίς να φτάσουμε έως εκεί θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε προς μια πολιτική που να μπορεί να ανοίξει την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας στις απαραίτητες πηγές πρωτογενούς ενέργειας για να έχουμε ανεφοδιασμό και κατανάλωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική συζήτηση στην Ευρώπη και πρέπει να γίνει. Έχουμε λάβει ήδη θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ σε εφαρμογή ορισμένα είναι πολιτική ανταγωνισμού και εργαλεία. Το τρίτο πούμε νομοθετικό πακέτο για την ενέργεια που εγκρίθηκε στα τέλη της προηγούμενης θητείας εν μέρη βασίζεται στην έρευνα που κάναμε στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο. Θα πρέπει να προχωρήσουν οι διασυνδέσεις, θα πρέπει να προχωρήσουν οι στόχοι κατά πολέμησης κλιματικής αλλαγής που θα μας οδηγήσουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης κλπ. λοιπά, Πάει λέγοντας. Είναι πολλά όμως αυτά που πρέπει να γίνουν. Ε, υπάρχουν και εργαλεία και ανταγωνισμού που μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν, αλλά δεν είναι αποκλειστικά ανταγωνισμού, ούτε τα σημαντικότερα είναι στον ανταγωνισμό. Το ζήτημα είναι πολιτικό και κεφαλαιόδου σημασίας. Στη συνέχεια, σε σχέση με τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε στη διακομματική ομάδα στο Intergroup για τις κοινοφελείς υπηρεσίες, πολύ ενδιαφέρον ε, ήταν. Σας είπα, δεν έχουμε αποκρισταλώσει θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς το άρθρο 14 της συνθήκης ερμηνεύεται και αναπτύσσεται. Όταν ήρθε ο πρόεδρος Μπαρόσο στο Κοινοβούλιο, για να τον επιβεβαιώσετε ως Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ξέρω τεχνικά πώς το λέτε, πριν διοριστεί και αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέρσι το Σεπτέμβριο δώσατε ψήφο εμπιστοσύνη. μίλησε για ένα ποιοτικό πλαίσιο. Ο καθηγητής Μόντι στην έκθεσή του για την εσωτερική αγορά μιλεί για τη δυνατότητα να αναπτυχθεί το άρθρο 14 μέσω κανονισμών, όπως άλλωστε και το ίδιο το άρθρο 14. Δηλαδή, να έχετε υπόψη ότι μπορεί να αποβεί πιο εύκολο ε, με κλαδική αντιμετώπιση. Και υπάρχουν τέτοιε ήδη στι τηλεπικοινωνίε, στο ταχυδρομείο, στι μεταφορέ. Παρά να υπάρχει μια οριζόντια έτσι, ε, μορφή κανονισμού. Πάντω το θέμα εκκρεμεί ακόμα, θα το συζητήσουμε, θα το σκεφτούμε και εν ευθέτω χρόνο θα αποφασίσουμε. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι δύο είναι οι σαφείς αρχέ Στη συνθήκη της Λισαβόνας και πριν την αρχή της Λισαβόνας και αφορούν άμεσα τον ανταγωνισμό. Ότι η πολιτική ανταγωνισμού δεν έχει κανένα λόγο να περιορίζεται λόγω μεγέθους. Μπορεί να υπάρχει υποχρέωση κοινοποίηση ή όχι μια κρατική ενίσχυση. Αλλά τα κριτήρια για το κατά πόσο χορηγείται μια κρατική ενίσχυση και είναι συμβατή ή όχι, δεν θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθο εκείνου που βοηθά. Και το δεύτερο, πάντα μιλώντα για κοινοβουλίες υπηρεσίε και γενικού συμφέροντος, είναι μια αρχή αναγνωρισμένη ρητά από τη συνθήκη, που είναι αρχή τη διαφορετικότητα. Διαφοροποίηση. Δεν θα πρέπει από εδώ και δεν επιτρέπεται εμείς να επιβάλλουμε τον ορισμό. Τι είναι κοινοφελή υπηρεσία σε κάθε χώρα. Ούτε λογικό είναι, ούτε θα το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ούτε και θα το δεχθούν. Ούτε τα θεσμικά όργανα και οι θεσμοί δημοκρατικοί της κάθε χώρας. Σε κάθε χώρα έχουμε διαφορετικά οράματα, κριτήρια, παραδόσεις. Μπορεί να μοιραζόμαστε κοινέ αξίες και κοινέ φιλοδοξίες, δεν λέω. Αλλά ένας ευρωπαϊκός κανονισμός δεν μπορεί να είναι, ε, ούτε επιτρέπεται ασύμβατος με τη διαφορετικότητα. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, Εμείς θα κάνουμε εκείνο που μας αναλογεί για να έχουμε γενικά πολύ καλές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, το άρθρο 106, τις συνθήκες. Θα δούμε και το άρθρο 14 πώς θα αναπτυχθεί, πώς θα εξελιχθεί, πώς το πρωτόκολλο 27 θα ερμηνευθεί η βάση του άρθρου 14, αλλά το ε, άρθρο 106 πρώην 86 ε, ήταν, είναι και θα είναι σε ισχύ και θα το εφαρμόζουμε κάθε μέρα. Τελευταίο, αυτό που με ρώτησε η κυρία Κράτσα. σε γερμανικό περιοδικό έδωσα αυτή τη συνέντευξη στην οποία αναφερθήκατε. Εγώ γερμανικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι διαβάσατε εσεί εσείς σε αυτή την εφημερίδα. Ξέρω όμως τι είπα και ξέρω τι μετέφρασαν και τι έγραψε το περιοδικό, η εφημερίδα, συγγνώμη. Και σε αυτή τη συνέντευξη μίλησα για ισπανικέ και ελληνικέ τράπεζε, αλλά ήθελα να πω το εξή. Όπω οι βρετανικέ τράπεζε, οι ιρλανδικέ τράπεζε, οι γερμανικέ, οι βελγικέ, οι ολλανδικέ, θα μπορούσα να σα αναφέρω κι άλλε. Ήδη έχουν λάβει πολλέ ενισχύσει, ε, αύξηση κεφαλαίου. Στην περίπτωση τη Ελλάδα, ακόμα η διαδικασία αυτή δεν έχει λάβει χώρα. Ενδεχομένω θα πρέπει να το σκεφτούμε, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα Υπήρξαν προγράμματα ρευστότητα, αλλά όχι αύξηση κεφαλαίου. Ούτε έγινε πολύ μεγάλη χρήση κρατικών εγγύσεων, γιατί βρήκαν από άλλους δρόμους και διάβλου ρευστότητα. Και στην περίπτωση τη Ισπανίας τώρα μόνο αρχίζουν να θέτουν σε εφαρμογή τις δύο μοναδικές αποφάσεις που ελήφθησαν για ενίσχυση κεφαλαϊκή ε, για δύο μικρά ταμιευτήρια. Αυτό λοιπόν δεν είναι συνώνυμο σε αύξηση κεφαλαίου γιατί ε, ήδη έχει δημοσιευθεί ο κατάλογος ποιος θα πάρει ε, χρήματα από τον οργανισμό αυτό τον Ισπανικό όταν εγκριθεί από την Ισπανία. Δηλαδή μιλούσα για χρονική καθυστέρηση, για διαφορά φάσεως. Ε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες χώρες, αλλά η Ισπανία και η Ελλάδα δέχτηκαν, επελήγησαν από την χρηματοοικονομική κρίση αργότερα από άλλες χώρες. Αυτό μπορεί να είναι καλό ή κακό. Καταρχήν μπορεί να φαίνεται καλό. Γιατί στην αρχή οι τράπεζές τους δεν επλήγησαν τόσο πολύ. Ε, όσο διαιωνίστηκε η κρίση έφτασε και εκεί και έφτασε και στην Ελλάδα συγκεκριμένα και γνωρίζουμε ότι έφτασε και από άλλα κανάλια που ε, επηρεάζουν και το χρηματοοικονομικό σύστημα και το χρηματοπιστωτικό. Εν πάση περιπτώσει, η ενίσχυση ε, της Ελλάδας για το δημόσιο χρέος, τα 110 δις που ενέκνε το Συμβούλιο, έχει και ένα υποκεφάλαιο 10 δις που πηγαίνουν σε ένα ταμείο σταθεροποίηση για ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Αυτό ήθελα να σας πω. Και το λέω στα ισπανικά πιο σαφώς από ό,τι στα γερμανικά. Stress and competition. un ejercicio. Το stress test έχει να κάνει με όλα. Δεν, ξέρω αν είναι ανταγωνισμός μπορεί να έχει να κάνει με ανταγωνισμό εξαρτάται, θα δούμε, θα δημοσιευθούν τα stress test και αν χρειαστεί ενίσχυση κεφαλαίου κάποια τράπεζας, αυτή μπορεί να γίνει ίσως ε, μέσω των αγορών με αύξηση κεφαλαίου ή αν δεν βρεθούν ε, ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει ε, κάποιος δημόσιος επενδυτής να είναι και αυτή τη στιγμή θα μπούμε σε δράση από πλευράς ελέγχου δηλαδή των κρατικών ενισχύσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Επίτροπο. Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας. Την ε, Δευτέρα στις 28 ε, Ιουνίου θα είναι η επόμενη συνεδρίασή μας. Την επόμενη Δευτέρα δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ.